Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε τώρα τη συζήτησή μας. Τώρα έχουμε τα Δυτικά Βαλκάνια, Δήλωσε της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής ΥΠΑ της Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικά Βαλκάνια. Για να ξεκινήσουμε θα παρακαλέσω την Αντιπρόεδρο κυρία Μογκερίνη να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ.